Λοιπόν κυρίε και κύριοι, τα πρακτικά της τη 24 24η έκτου έχουν ε, ήδη γνωστοποιηθεί. Υπάρχουν ενστάσεις, δεν υπάρχουν. Κυρώνονται τα πρακτικά. Κύριε Φερχόφστατ, ζητήσα τον λόγο για διαδικαστικό. Πρόεδρε, Θέλω να σας ευχαριστήσω για την στήριξη αυτή, τη δήλωση που μας απευθύνατε. Θέλω να υποφεληθώ πάντως από αυτή την ευκαιρία, ώστε εκ μέρου του Άλτε και 152 σημείο 1 να σας πω το εξή. Προσπαθούμε να εγκρίνουμε ψήφισμα, ένα ενιαίο ψήφισμα για την Σρεμπρένιτσα. Γι' αυτό και προτείνω αυτό να γίνει την Πέμπτη το πρωί. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε και το ψήφισμα αυτό με το οποίο θα τιμήσουμε τα θύματα της Ρεμπρένιτσα. Θα τιμήσουμε συγχρόνως και όλα τα θύματα από τον πόλεμο στην τέος Γιουγκοσλαβία και θα ανοίξουμε μια νέα προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια, όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, στην ομιλία σας. Το χρειαζόμαστε το ψήφισμα αυτό. Ο κόσμος μας χρειάζεται μια τέτοια δήλωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας προτείνω όταν στη συνέχεια περάσουμε στα θέματα της Πέμπτης να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Θα σας δώσω τον λόγο τότε στη συνέχεια. Εντάξει. Κύριε Χάνς, ζητήσατε τον λόγο για διαδικαστικό. Η κυρία Ρεμπέκα Χάνς, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, αυτή την εβδομάδα με σαφήνεια θα καθοριστεί σε σχέση με τις συζητήσεις που αφορούν το δημοψήφισμα στην Ελλάδα και νομίζω ότι η Ελλάδα σε εμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά που βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ε, απευθύνεται σε εμά και αυτό οδηγεί στο ότι οι συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεδομένων μιας, ε, δεδομένης μιας τέτοιας εξέλιξης είχε προϋπάρξει κάποια προαναγγελία μπορεί να διαβάσει κανείς τα σχετικά ο Μάρτιν Σούλτς ως ε, πρώην αρχηγός της ε, πολιτικής ομάδας και ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου μπορεί να διαβάσει κανείς τι είπε τότε για να αποφευθεί αυτή η κατάσταση τι είναι τώρα σωστό τι είναι σωστό και τι είναι λάθος πλέον εγώ πιστεύω ότι ο πιο σημαντικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι που είναι το σώμα που είναι άμεσα έχει εκλεγεί από τους πολίτες της Ευρώπης από το Βορρά και το Νότο και την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη ρόλος είναι να δημιουργούμε γέφυρες που θα δημιουργούν διέξοδο από την κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να σας πω κύριε Σούλς και δεν είναι εύκολο να σας το πω αυτό επειδή το, ο πέμπτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είχατε μεγάλες ελπίδες από πλευράς μας Πιστεύω ότι η ομάδα μου έχει δίκιο. Έχει δίκιο η ομάδα μου. Ο τρόπος με τον οποίο εσείς ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμειχθήκατε στη συζήτηση για την Ελλάδα ήταν λανθασμένος, ανεύθυνος. Και αυτό όχι επειδή υποστηρίξατε το ναι στο δημοψήφισμα, όχι επειδή υποστηρίξατε το ναι στο δημοψήφισμα στην Ελλάδα, αλλά, αλλά, επειδή οδηγηθήκατε στην λανθασμένη τοποθέτηση και την αντιμετώπιση με τοπική που μεταξύ Ελλάδας και των άλλων χωρών είχε συμβεί συνεισφέρατε σε αυτή την υπόθεση και θέλω εδώ να σας πω ότι δεν είσαστε ενδεδειγμένος κύριε Σούλτς να αναλαμβάνετε ένα ενεργό ρόλο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή την οξύτατη φορτισμένη διαδικασία και θέλω να σας ζητήσω επιτέλους να απόσχετε, να αποστασιοποιηθείτε διότι η ζημιά που προκαλέσατε εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολύ μεγαλύτερη από το όφελος το οποίο δημιουργήθηκε, προκλήθηκε. Υποθέτω κυρία Σίμα στο ίδιο θέμα θέλετε κι εσείς να τοποθετηθείτε. Να τοποθετηθείτε. Σωστή υπόθεσή σας. Δεν ανήκουν πολλά να πει κανεί σε αυτά τα πράγματα και στην, την προηγούμενη εβδομάδα ο Δημήτρη Παπαδημούλη ω αντιπρόεδρο και εγώ ω πρόεδρο ε, τη Ενωτική Αριστερά αποστήλαμε ήδη επιστολή και διαμαρτυρηθήκαμε κατά τη κατάσταση αυτή. Ότι στην αρχή τη προηγούμενη εβδομάδα εσεί ενεργά ω πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκήσατε την επιρροή σα, αναμειχθήκατε στην διεξαγωγή του δημοψηφίσματο στην Ελλάδα. Εμεί πιστεύουμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μόνου αιρετού, άμεσα αιρετού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια δημοκρατική διαδικασία να αναμειγνύεται με αυτόν τον τρόπο σε ένα κράτος μέλος. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Ούτε όταν πρόκειται για το δημοψήφισμα στη Σκωτία, ούτε στα δημοψηφίσματα στην Ολλανδία, εντάξει τότε δεν είσαστε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ομολογώ, αλλά και σε άλλα δημοψηφίσματα. Ποτέ δεν είδαμε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προαναγγέλει μια εκστρατεία που ξεκινά και να λέει ότι πρόκειται να αναμειχθεί για ένα ναι σε ένα δημοψήφισμα, σε μια εκστρατεία και ταυτόχρονα λέει ότι μια κυβέρνηση την διαδρομή της και έχει τερματίσει τη διαδρομή της και πρέπει να ακολουθήσει μια τεχνική λέει κυβέρνηση τεχνοκρατών. Και ταυτόχρονα ταυτόχρονα για έναν εκλεγμένο πρόεδρο να λέτε ότι είναι ένας δημαγωγός είπατε και νομίζω ότι δεν έχει καμιά σχέση αυτό τέτοιες δηλώσεις ε, με τη δική σας ιδιότητα ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία και σε αυτήν είχατε αναμειχθεί και προσπαθήσατε λέει να δυναμώσετε τα δικαιώματα ενδυναμώσετε τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όμως δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι είσαστε εσείς το Κοινοβούλιο δεν είσαστε εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εσείς λάβατε εντολή από εμάς ως πρόεδρος. Και δεν λάβατε όμως την εντολή να κάνετε τέτοιες δηλώσεις και τέτοιες τοποθετήσεις. Παρακαλώ στο μέλλον να απόσχετε και να αποστασιοποιηθείτε από τέτοιου είδους πράξεις. Κάθε λαός έχει το δικαίωμα σε ένα δημοψήφισμα σημαντικές υποθέσεις που αφορούν αυτό το λαό να τις ρυθμίζει με τον τρόπο που κρίνει ότι είναι σωστός. Και για ένα ερετό δημοκρατικό σώμα που είσαστε εσείς πρόεδρος του έχετε το καθήκον να προασπίζεστε τη δημοκρατία εξ ονόματός του. Δεν είναι δυνατόν ε, να είναι η πιο αδύναμη κρίκη της αλυσίδας ε, η εκλογής. Ε, πρέπει να συζητηθούν εναλλακτικέ λύσεις και να ψηφιστούν. Σας ζητώ κατεπηγόντως ακριβώς αυτή την πρόταση να υιοθετήσετε και υπό το δικό μας πρίσμα πρέπει να ξαναβρείτε τη σωστή πορεία κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, τώρα φυσικά πάρα πολλές παρεμβάσεις ε, έλαβαν χώρα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση γιατί σύμφωνα με τον κανονισμό συζητήσεις για τέτοιου είδους θέματα δεν είναι δυνατόν να διακόπτονται. Πήρατε και περισσότερο χρόνο από ότι ανήκει σε μια παρέμβαση επιδιαδικαστικού Και θα πρέπει να σκεφτείτε, θέλετε να διεξαχθεί τώρα συζήτηση επ' αυτού, εδώ στην Ολομέλεια. Κάπως με εκπλήσει όταν πρόκειται για την Ουγγρική κυβέρνηση μου ζητούν με, όλα τα, με όλες τις δυνάμεις μου να εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναντί της Ουγγρικής κυβερνήσεως. Εγώ δεν ζήτησα η ελληνική κυβέρνηση να αποπεμφθεί, να διαβάζετε ακριβώς τα κείμενα προτού φωνάζετε εδώ στην Ολομέλεια. Να το σκεφτείτε λοιπόν σε βάθος αν θέλετε να εμβαθύνετε σε αυτή την υπόθεση με συζήτηση κυρίες και κύριοι. Ξαναρωτώ, παρακαλώ κύριε Φεχόφστατ. Uh, Έχω ένα θέμα για τη συζήτηση της Τετάρτης. Τώρα να αναφερθώ σε αυτό. Μάλιστα, θα το κάνουμε αμέσως, θα το ρυθμίσουμε αμέσως. Oh, Την Τετάρτη, για τη συζήτηση στην Ελλάδα. Θα περάσουμε αμέσω τώρα στην ημερήσια διάταξη. Θα περάσουμε αμέσω στη συνέχεια στην ημερήσια διάταξη και θα παρέμβετε. Θέλει κάποιο άλλο να παρέμβει, παρακαλώ. Όχι, δεν θέλει κανεί. Ευχαριστώ λοιπόν. Παρακαλώ κύριε Πιτέλα. Παρακαλώ. Εγώ κύριε Πρόεδρε δεν θεωρώ ότι όταν εκλέγεται κάποιος πρόεδρος του Κοινοβουλίου χάνει το δικαίωμα στην άποψή του. Και πρέπει να πω με πάσα ειλικρίνεια ότι όταν ε, συναντήθηκα με τον Μάρτιν Σούλτ πριν από κάποιους μήνες ε, και δημοσίως και ιδιωτικώς Άκουσα πάντα τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Μάρτιν Σούλτ, που είναι και σύντροφό μου στην ομάδα, να λέει ε, πράγματα τα οποία ήταν υπέρ τη συνεργασία προ εξέβρεση λύση, ώστε να επιτραπεί η διάσωση της Ελλάδος και η συγκεκριμένη εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους Έλληνες πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι είναι σφάλμα σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για την ε, ιστορία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων να επινοούμε στόχους που δεν είναι οι σωστοί στόχοι. Θα πρέπει αντίθετα να επικεντρωθούμε στο τι πρέπει να γίνει προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη και η Ελλάδα να διαφύγουν από αυτή τη ε, στιγμή εξαιρετική δυσκολίας. Εγώ επιβεβαιώνω τη δέσμευση τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει προκειμένου να σώσει την Ελλάδα. Ε, σεβόμενοι και τα ε, υποχρεώσεις της ελληνικής κυβέρνησης και σεβόμενοι και την αλληλεγγύη που πρέπει να επιδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να ε, ξεκινάμε φιλονικίες ενώπιον ενός ανθρώπου, ο οποίος στη διάρκεια της προεδρίας του έφερε στο πιο υψηλό επίπεδο την εξουσία, το κύρος και την, ε, και την κυριαρχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ζητούν άλλοι τον λόγο πλέον σε σχέση τώρα με την παρέτηση του κ.